Και θα ήθελα τώρα να σας ε, ανακοινώσω ότι υπάρχει πρόταση ε, ψηφίσματος. Και έτσι λοιπόν κλείνει η συζήτηση. Ε, θα ψηφίσουμε αύριο στις 12 ε, το μεσημέρι. Το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι μια έκθεση του κυρίου Βόγκαν. πρόκειται για τις κατευθυντήριες γραμμές για τον προεπολογισμό του 2013. Πρώτος ομιλητής είναι ο εισηγητή. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Κύριος Μπόουν. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρε, δεν είναι εύκολο να καθορίσει κανείς τον προπολογισμό του, οπότε θα πρέπει να ξεκινήσω ευχαριστώντας όλους τους Η εισηγητάς, το Προεδρείο και τον Γενικό Γραμματέα για την αγαστή συνεργασία που είχαμε όσον αφορά την εκπόνηση αυτών των κατευθυντηρίων. Νομίζω ότι έχει διαμορφωθεί μια ευρεία συνένεση. Όμω, μια που είμαστε μια δύσκολη συγκυρία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να διαδραματίσει τον ρόλο του και θα πρέπει να προβεί σε περικοπέ. Επίση, θεωρώ ότι πάρα πολύ λίγοι θα διαφωνούσαν ε, με το πάγωμα του προπολογισμού που προτείνουμε. Άρα θα πρέπει να έχουμε αύξηση κάτω από τον προϋπολογισμό. Δεν συζητιέται επομένω το ότι υπάρχει ο πληθυσμό, όμω υπάρχει ευρεία συμφωνία, ευρεία είναι σχετικά με αυτό. Έχουμε επομένω αυτέ τι συστάσει για τι καθηγητήρε, οι οποίε νομίζω ότι έχουν γίνει αποδεκτέ και είναι πάρα πολύ σημαντικό ω κοινοβούλιο να μπορέσουμε να επισημάνουμε, να βρούμε, να βάλουμε κάποιε περικοπέ στον προπολογισμό και να κάνουμε δαπάνε μόνο δεν είναι απολύτω αναγκαίε. Θεωρώ επομένω ότι θα πρέπει να παγώσουμε τα οδηπορικά ε, γιατί το, το ζήτησε αυτό και ο Γενικός Γραμματέας. Άρα, να παγώσουμε όλα τα σχετικά επιδόματα προς τους βουλευτές, ε, την μέση αποζημίωση, την αποζημίωση για το γραφείο, όλα αυτά να παγώσουν, να παγώσουν μέχρι το τέλος αυτής της θητείας. Επίσης να κάτσουμε και να ξαναδούμε όλα τα κονδύλια, κυρίως τα κονδύλια εκείνα τα οποία ε, συνήθω δεν βρίσκονται σε υποαπορρόφηση. Και έτσι να πετύχουμε τις οικονομίες που χρειαζόμαστε επομένως να εξασφαλίσουμε το ότι έτσι θα μπορέσουμε να καλύψουμε οτιδήποτε προκύψει σε σχέση με τα κτίρια. Στο παρελθόν είχαμε ένα σωρό προτάσει για κτίρια, Όλα αυτά τώρα τα λάβουμε υπόψη. Χρειαζόμαστε διαφάνεια. Διαφάνεια και έτσι θα πρέπει το Κοινοβούλιο να ενημερώνεται για τα οράματα, τα σχέδια που υπάρχουν, τι προτάσεις για κτίρια. Και αυτό να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Άλλη πρόταση. Περισσότερη συνεργασία μεταξύ των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων. Κτίρια. Διερμηνία ανθρώπινη πόρη. Ε, να συνεργαστούμε με την Επιτροπή των Περιφερειών και με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή για όλα αυτά τα θέματα. Ίσως θα πρέπει επομένω να δούμε τι κοινή συμφωνία μπορεί να υπάρξει σε σχέση με τις παλαιότερες από τις οποίες μπορούμε να αντιλήσουμε συμπεράσματα και επομένω έτσι μπορούμε να κάνουμε οικονομίες. Υπάρχει, υπάρχει περιθώριο και στην μετάφραση. Επομένω, θα, θα, θα, κάτσουμε και θα δούμε πού μπορούμε να κάνουμε εξοικονόμηση δαπανών. Και ο, ο, ο κύριος Γενικός Γραμματέα πρόκειται να κατεβάσει προτάσει για το πώ θα έχουμε μια ανεξάρτητη αξιολόγηση των πραγμάτων για τον προπολογισμό και έτσι θα έχουμε ένα φρέσκο βλέμμα πάνω στον προπολογισμό. Επομένω, αυτό σα ε, προτείνω να συγκροτήσουμε ομάδα εργασία. Ε, η Επιτροπή των Προπολογισμών και το Προεδρείο να κάτσουν να φτιάξουν αυτήν την ομάδα και έτσι να δούμε τι οικονομίες μπορούμε να κάνουμε και έτσι να έχουμε αυτή την ανεξάρτητη αξιολόγηση του προπολογισμού μας. Επίσης, να κάνουμε συγκριτική μελέτη. Επί τη βάση της φετινής χρήσης, μία σύγκριση με άλλα κοινοβούλια στην Ευρώπη, αλλιώς και με το Αμερικανικό Κογκρέσο. Επίσης, να δούμε και τα οδηπορικά. Και φέτος θα γίνει κάποια έκθεση για τα φετινά, είπαμε, για τα δύο όλα αυτά ομάδα εργασία. Τέλος, συνάδελφοι. Προβληματίζομαι όσον αφορά τα του παγώματος. Και εγώ και οι άλλοι συνάδελφοι και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όμως, άλλοι θέλουν να προχωρήσουμε ακόμα πιο μακριά και να περικόψουμε κονδύλια. Έχουμε και τέτοιες τροπολογίες τις οποίες θα ψηφίσουμε αύριο. Οι περισσότεροι συνάδελφοι θα συμφωνούσαν ότι τελικά θα καταλήξουμε σε ένα σύμβασμο. Αυτός είναι ο δρόμος. Αυτό είναι η κατεύθυνση που θέλουμε να πάρουμε και έτσι να μπορέσουμε να έχουμε έναν υγιή προϋπολογισμό αλλά ταυτόχρονα να έχουμε και εύρυθμη λειτουργία του Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστούμε για την εισήγησή σας, λέει ο Πρόεδρος. Τώρα, κύριε Χολμάγερ, για τρία λεπτά. Αξιότιμε πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα ξεκινώντας να ευχαριστήσω τον ε, συνεισηγητή τον κύριο Βόν για τη θαυμάσια συνεργασία και για την ε, προθυμία του να εξετάσουμε σε βάθος όλα τα θέματα και να αναζητήσουμε λύση. Ήδη πέρυσι καταθέσαμε ε, προπολογισμό λιτότητας ε, όπου ο αρχικός προϋπολογισμός αυξήθηκε κατά μόνο 0,8% και το επιπρόσθετο κόστος με την διεύρυνση με την ένταξη της ε, Κροατίας ε, συγκρατήθηκε και παραμείναμε στην αύξηση του μόνο 1,9%. Και φέτος λοιπόν ε, θέλουμε να έχουμε προπολογισμό λιτότητας και με τον τρόπο αυτό να αποδείξουμε ότι γνωρίζουμε ότι βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον όπου δεν μπορεί κανείς να προβεί σε χρηματοδοτικά ή χρηματοψηφιακά άλματα. Αυτό που θα πρέπει να έχουμε κυρίως κατά νου είναι η δημοσιονομική αποτελεσματικότητα. Χαιρετίζω την ε, σύσταση ομάδας εργασίας η οποία ακριβώς θα έχει ως στόχο από κοινού με το Προεδρείο, τη Γραμματεία και τη Διοίκηση του Προπολογισμού να καταβληθούν προσπάθειες για να καταφεύγουμε σε εξωτερικούς εμπειρογνώμονες μόνο εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι απαραίτητο να ενισχύσουμε περαιτέρω τη θεσμική συνεργασία και επίσης ε, να ε, μεριμνήσουμε ε, έτσι ώστε οργανωτικά το Κοινοβούλιο να είναι αποτελεσματικό να βελτιστοποιήσουμε περαιτέρω τη χρήση του προσωπικού. Και γι' αυτό το λόγο πέρυσι, παραδείγματος χάρη, και μόνο στον τομέα της μετάφρασης και της διερμηνίας, μέσα σε ένα χρόνο εξοικονομήσαμε 21 εκατομμύρια ευρώ και αυτό επιθυμούμε να πράξουμε και φέτος. Όπως είπε και ο συνάδελφος κύριος Βον, έχουμε παγώσει τις δαπάνες ταξιδίου και τις αποζημιώσεις, τις ημερήσεις αποζημιώσεις και όσον αφορά την πολιτική ακινήτων, εγώ είμαι συγγήτρια για αυτήν την πολιτική, θεωρώ ότι πρέπει να εξετάσουμε το κατά πόσον η πολιτική ακινήτων, ε, κυρίως ε, τα ε, προγράμματα ανέγερσης νέων κτηρίων, κατά πόσον αυτά εφαρμόζονται αποτελεσματικά έτσι ώστε να εξοικονομούνται δαπάνες, κυρίως σε ετήσια βάση. Σημασία έχει να χρησιμοποιούμε συνέργειες. Περιμένουμε και από άλλους θεσμούς να συμφωνήσουν μαζί μας, να μας στηρίξουν. Θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να ακολουθήσουμε έναν δρόμο όπου αφενός ε, το Κοινοβούλιο θα εργάζεται με ακρίβεια και πολύ συγκεκριμένα, από την άλλη όμως θα είναι και αποτελεσματικό. Ευχαριστώ το Προεδρείο, τη Γραμματεία ε, για την πολύ καλή συνεργασία και εύχομαι να επιτύχουμε έναν ε, σταθερό, καλό προϋπολογισμό. Ευχαριστούμε κυρία Χούλμαια και για δύο λεπτά η κυρία Χάτσουκ. Αγαπητοί συνάδελφοι, επιτρέψτε μου ε, καταρχήν να συγχαρώ τον κύριο Ντέρκ Βόν, ο οποίος ε, ε, προετοίμασε και συντόνισε τις εργασίες για την έκθεση. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό ο προϋπολογισμός του 2010 να παρουσιάσει ουσιαστικά αποτελέσματα, κυρίως προς την κατεύθυνση της εξοικονόμησης. Αυτό που μας ενδιαφέρει να υπάρχει σωστή διαχείριση ε, και στους ε, άλλους κοινωτικούς θεσμούς εκτός ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ένωσης. Κυρίως πρέπει να ξεκινήσουμε εδώ, σε εμά με την εξοικονόμηση. Γιατί όχι στους βουλευτές. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό να παγώσουν οι μερίσεις αποζημιώσει, ε, να περιοριστούν οι δαπάνε ταξιδίου, να περιοριστεί ε, και το κόστος της μετάφρασης. Παράλληλα είναι πολύ σημαντικό να μην προχωρήσουμε σαν οδοστρωτήρα. Πρέπει να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα. Είναι σημαντικό όχι μόνο να ε, εξοικονομούμε χρήματα αλλά και να επενδύουμε. Ε, χρειαζόμαστε την τεχνική, ε, τεχνολογική καινοτομία. Αυτό είναι σημαντικό αν θέλουμε να εργαζόμαστε με καινοτόμο τρόπο. Όσον αφορά την ένταξη της ε, Κροατίας, οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι εκεί δεν μπορούμε να εξοικονομήσουμε χρήματα. Οι, εργα... οι ε, βουλευτές από την Κροατία, οι συνεργάτες από την Κροατία έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα με εμά. Γι' αυτό λοιπόν ε, θα πρέπει να επιδείξουμε κάποια διαφοροποίηση. Και θέλω να επισημάνω ότι το κόστος για τους συνεργάτες, αν επιθυμούμε να περιορίσουμε αυτό το κόστος, οφείλουμε να έρθουμε σε διαβουλεύσεις με, τους, ε, με τα συνδικάτα. Και εγώ προσωπικά χαίρομαι πάρα πολύ που θα συσταθεί μια επιτροπή στην οποία θα συμμετέχει το Κοινοβούλιο, η Γενική Γραμματεία, η Επιτροπή Προϋπολογισμών και αυτή η ομάδα εργασίας θα επιληφθεί της ε, πολιτικής ε, λιτότητας. Ευχαριστώ όλους όσοι συμμετείχαν στις μέχρι τώρα εργασίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ότι τηρήσατε το χρόνο σας και το ε, λόγο έχει τώρα ο συνάδελφος ε, Γκεμπράντι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον Τέρεκ Βόν για το εξαιρετικό του έργο και για τον πολύ ευχάριστο τρόπο με τον οποίο μπόρεσε να συνεργαστεί με τους και Ευχαριστώ λοιπόν οι προηγούμενοι δύο ομιλητές για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες και το ΕΛΚ έδειξαν ότι κάτι κινείται στο σώμα αυτό, ιδίω ω προ το θέμα του προπολογισμού. Ήταν πολύ δύσκολο να κάνουμε οικονομίε και ιδίω πέρυσι. Βλέπω όμω τώρα ότι το σύνολο του Κοινοβουλίου είναι πλέον προετοιμασμένο για να δει με τρόπο αρκετά κριτικό την ίδια του την διαχείριση. Η οικονομική κρίση εμένει. Αυτό σημαίνει ότι θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες εξοικονόμησης κονδυλίων. Μόνο μία πραγματική απάντηση υπάρχει εδώ. Χρειαζόμαστε πολύ περισσότερη διαφάνεια. Και εδώ έχουμε έναν τομέα όπου απαιτείται περισσότερη δουλειά από μέρους μας. Εδώ πρέπει να διερευνήσουμε τον ίδιο μας τον προπολογισμό και να δούμε πώς θα ε, κάνουμε ακόμη περισσότερες οικονομίες στο Κοινοβούλιο. Πέρυσι η Ολομέλεια τα αντιμετώπισε αυτά με την αφορμή της έκθεσης απαλλαγής. Δυστυχώς το Προεδρείο δεν αντέδρασε θετικά. Ο κύριος Φερχόφστα τον ε, Δεκέμβριο μόλις απέστειλε επιστολή στον Πρόεδρο Μπούζεκ και το θέμα αυτό γιατί ζητούσε να γίνουν, ε, να ληφθούν, να ληφθεί ανάλογη μέρημνα για τον προπολογισμό θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω, Πρόεδρε, να λάβετε υπόψη σοβαρά το θέμα αυτό. Χρειάζεται να αναθεωρήσουμε όλες τις γραμμές του προπολογισμού και να υπάρχει σωστή επιλογή. Η Επιτροπή Προπολογισμών θα μπορούσε έπειτα να εξετάζει την ε, μελέτη αυτή προκειμένου να δούμε πού μπορεί να γίνουν οικονομίες. Συμφωνούμε ότι οι γενικές γραμμές για το πάγωμα των δημοσιονομικών γραμμών είναι σωστές και θα πρέπει να έχουμε έναν ακόμη πιο λιτό προπολογισμό για το σώμα μας φέτος. Ευχαριστώ να δώσω το λόγο στον κύριο Άσπροθ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Προεδρεθνικές κυβερνήσεις σε όλη την Ευρώπη καταβάλουν προσπάθειες για να περικόψουν τις δαπάνες και να ε, κάνουν τα κονδύλια αποτελεσματικά, καθώς και να ελέγχουν αυστηρά τους προπολογισμού τους. Αυτό είναι και δική μας δουλειά. Ως μέλη του Κοινοβουλίου πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε το ίδιο. Πρέπει στενά να παρακολουθούμε τους προπολογισμού του σώματό μας και να επιβάλλουμε αυστηρότητα στον έλεγχο. Εδώ έχουμε μια πραγματική ευκαιρία να δείξουμε ότι μπορούμε να έχουμε πρωταγωνιστικό ρόλο. Θα πρέπει εδώ να αποτύσσω φόρο τιμή στο Γενικό Γραμματέα και το Προεδρείο του Κοινοβουλίου για τα πολύ ρεαλιστικά στοιχεία και τι προτάσει που μα υποβάλλουν σήμερα. Όμω θέλω ταυτόχρονα να πω ότι Πρέπει να διερωτηθούμε αν έχουμε το δικαίωμα ω μέλη αυτού του σώματο να απαιτούμε από άλλα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση να ακολουθούν το παράδειγμά μα. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να απαιτούμε πραγματικέ οικονομίε και στου δικού του προπολογισμού και ότι εκείνοι θα οφείλουν να αποδεικνύουν ότι και οι δικέ του δαπάνε είναι αποτελεσματικέ. Εδώ λοιπόν στηρίζω πλέον πλήρω την ε, παρέμβαση του εισηγητή για περισσότερε οικονομίε και σε πολλού τομεί θα μπορούσαμε να πάμε ακόμη παραπέρα. Για την ώρα πάντω συγχαίρω τον για την εξαιρετική του. Ωστόσο, Υπάρχουν τρία σημεία στα οποία ήθελα να σταθώ. Πρώτον, η πολιτική των κτηρίων. Τα μέλη του σώματο αυτού θα έπρεπε να είναι πιο επικριτικά ω προ τι επενδύσει για τα κτίρια, τη διαχείριση των κτηρίων και τον έλεγχο του κόστου των κτηρίων. Ιδιαιτέρω θα έπρεπε να περιμένουμε και τα άλλα θεσμικά όργανα να επιτύχουν μεγαλύτερη αποδοτικότητα μεταξύ της κατανομή, μέσω μάλλον της κατανομής των πόρων. Δεύτερον, η διοίκηση και το κόστος του προσωπικού. Το Κοινοβούλιο θα έπρεπε να εξετάσει τις ε, δυνατότητες των θεσμικών οργάνων να κάνουν σταδιακές οικονομίες μέσω ελέγχου του προσωπικού. Θα πρέπει να δούμε και τι κατηγορίε του προσωπικού και το υπηρεσιακό του καταστατικό και την πολιτική για το προσωπικό, για να είναι και επίκαιρα και εύστοχα και βεβαίω να ε, είναι αποδοτικέ οι δαπάνε των Ευρωπαίων φορολογουμένων. Τρίτον, δεν θα πρέπει η συζήτηση αυτή να μην περιλαμβάνει και κάτι πολύ σημαντικό για το Κοινοβούλιο. Την έδρα μας εδώ θα πρέπει να σκεφτούμε ότι εφόσον εγκρίνουμε την έκθεση αυτή, αποδεχόμαστε ότι η έδρα του Κοινοβουλίου είναι κάτι που πρέπει να συζητηθεί περαιτέρω. Δεν μπορούμε εμεί να προωθούμε την εξοικονόμηση, τη μείωση του κόστου, την αποτελεσματικότητα για τα άλλα θεσμικά όργανα, για τι άλλε κυβερνήσει και να είμαστε μεταξύ αυτών τη Ευρώπη που δαπανούμε ε, άσκοπα ε, κονδύλια. Έτσι λοιπόν συστήνω και στον εισηγητή και στα μέλη του σώματο ότι προκειμένου να παραμείνουμε αξιόπιστοι ω κοινοβούλιο θα πρέπει τη συζήτηση για την έδρα μα να την κάνουμε και να την κάνουμε πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ. Και τώρα ο κύριος Πόρτας για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Οι γενικοί προσανατολισμοί για τον ερχόμενο προπολογισμό του Κοινοβουλίου αποδεικνύουν ότι υπάρχουν προσπάθειες, προσπάθειες ε, εγκράτειας που οδεύουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Όμως η Ολομέλεια φαίνεται να αποκλεί από τη συζήτηση και τις προφορίες μία πρόταση που έχω υποβάλει και την οποία θέλω να διαβάσω. να διαβάσω. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμφωνήσει με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να παγώσουν οι μισθοί των Ευρωβουλευτών στις αξίες και στις τιμές του 2012. Η πρόταση αυτή θεωρώ ότι είναι μετριοπαθής, λογική και δεν υπάρχει κανένας λόγος να αποκλείεται από τις συζητήσεις μας. δεν ε, ε, αφαιρούμε κάτι από τους μισθούς των βουλευτών, ούτε χρειάζεται να παρέμβουμε στο καθεστώς ε, το... που διέπει τα μέλη του σώματος στο Κοινοβούλιο. Θα έπρεπε να μπορούν να αποφανθούν τα μέλη του σώματος για τα ε, ίδια τα εισοδήματά του. Αυτό θα ήταν σημαντικό για την εικόνα που δίνουμε εκτός Κοινοβουλίου. Γιατί καμιά φορά με τέτοιου φίλους η Ευρώπη δεν χρειάζεται καν του εχθρού. Σας ευχαριστούμε. Η κυρία Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε μέσα στην κρίση που τώρα σοβεί και θέλουμε να επιβάλλουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση περικοπέ στα κράτη-μέλη. Εμεί εδώ το Κοινοβούλιο θέλουμε, θέλουμε τη αριθμική αναπροσαρμογή. Δεν μπορούμε καν να συμφωνήσουμε ποιο θα είναι το ποσοστό τη ΑΤΑ. Όμω ε, λέμε 1,9, λέμε 3%. Το θέμα είναι όμω ότι η γραφειοκρατία ήδη ε, αυτή τη στιγμή έχει φουσκώσει και θα πρέπει να την να, να, να τη βάλουμε να κάνει δίαιτα, θα πρέπει να την συγκρατήσουμε. Ε, λέμε εδώ πέρα ότι το κόστος είναι 2 εκατομμύρια λίρες ανα, ανα, ανα ευρωβουλευτή. 160% έχει αυξηθεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια το κόστος τη ε, της ζωής. Άρα θα πρέπει όλες αυτές οι δαπάνες να καταργηθούν. Έχουμε εδώ πέρα μια παράδοση πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ είναι το κόστος εδώ, έχουμε κόστος λειτουργίας πάνω από 11 εκατομμύρια ετησίω. είναι επομένω μια σπατάλη όπως και να το δει κανεί. επομένως θα πρέπει όλη αυτή η υπόθεση να εγκαταλειφθεί. Η δε... Η δε χρηματοδότηση έχει αυξηθεί 176% τα τελευταία τέσσερα χρόνια, οπότε όλα αυτά ε, είναι τα πολιτικά κόμματα τα οποία δεν χρειαζόμαστε εμείς. Ε, εκλεγόμαστε από τους εκλογείς μας και από εθνικά ψηφοδέλτια. Κύριε Πρόεδρε, ο Ντέβιτ Κάμερον θέλει να υπάρχει μια, ένα, ένα πάγωμα, όμως αυτό που χρειάζεται είναι σημαντική μείωση και γενικά όσον αφορά τουλάχιστον 10% μείωση. Γιατί αλλιώς, αλλιώς αυτό μόνο θα κάνουμε θα είναι να διασπαθήσουμε τα χρήματα των φορολογουμένων. Τώρα λοιπόν για 1,5 λεπτό, ε, κυρία Μπέρτμαν, κοιτάξτε, σε αυτή την δύσκολη περίοδο η ρεαλιστική προσέγγιση του συναδέλφου Βόν είναι πολύ σημαντική και τη στηρίζουμε. Γιατί είναι σαφές ότι θα πρέπει να παγώσουμε τα κονδύλια για τη διοίκηση, κυρίως σε μια χρονική περίοδο όπου όλοι οι πολίτε καλούνται να σφίξουν, όπως λέμε χαρακτηριστικά, τη ζώνη, το ζωνάρι. Ε, σε τομεί ε, όπω οργάνωση προσωπικού ή διαχείριση κτηρίων πρέπει να υπάρχει καλύτερη συνεργασία. Ε, βεβαίως και είναι απαραίτητο να υπάρχουν προσπάθειε ελιτότητα, αλλά υπάρχουν και τομείς ε, όπου τα πράγματα πρέπει να είναι διαφορετικά. Περιβάλλον. Εκεί χρειαζόμαστε αποτελεσματική πολιτική. Ακριβώ οι δικοί μα οργανισμοί πρέπει να αποτελούν πρότυπο για την Ευρώπη. Και δεύτερον, στον τομέα τη μετάφραση και των γλωσσικών υπηρεσιών. Ήδη πέρυσι κατεβλήθηκε υπήρξαν προσπάθειες εξοικονόμησης κονδυλίων. Αυτό μας δεν μπορεί να ε, προχωρήσει στο διηνεκές. Αναφέρεται ε, στο ε, κανονισμό του Κοινοβουλίου ότι οι πολίτες πρέπει να μπορούν να παρακολουθούν τις συζητήσεις στη γλώσσα τους. Η διαφάνεια στις δημοκρατικές διαδικασίες δεν μπορεί να κολλείεται από λιτότητα στα κονδύλια για τη διερμηνία και τη μετάφραση. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω όλους όσοι προσπάθησαν. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, το λόγο έχει τώρα για τρία λεπτά ο Σνάλφος Γκαρίγκα Πολέντο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο προϋπολογισμός είναι, κάνει κάποιους είναι κάτι, κάτι σαν κυκλικά με φαινόμενο για μας εδώ πέρα. Οπότε κάθε φορά συγκεκριτής εδώ στο Κοινοβούλιο προσπαθεί να βρει μια ισορροπία μεταξύ των θεμητών συμφερόντων των βουλευτών, το μεταξύ των ευαισθησιών των εκλογέων αλλά και των αναγκών τη διοίκησης. Συγκεκριμένα για το δικό μα τον προπολογισμό, τον ευρωπαϊκό. Αυτό το οποίο θέλω είναι να σα πω αρχίζοντα ότι λειτουργεί εύρυθμα και τα περισσότερα κεφάλαιά του επίσης έχουμε όλο ένα και περισσότερες αρμοδιότητες και όλο και περισσότερα κράτη-μέλη. Το δε πολύπλοκο πρόβλημα της πολυγλωσσίας έχουμε 700 και βουλευτές το οποίο θα πρέπει να υποστηρίζουμε τεχνικά επομένως υπάρχουν πάρα πολλές πάρα πολλοί λόγοι γιατί είναι εκεί που είναι ο προπολογισμό ο πλευρά ύψου οικονομικού. Και λέμε, ε, μήπω λοιπόν, εκτό από αναγκαίο ο προπολογισμό, λέμε, εάν είναι βέβαια και βιώσιμο πρόθεσμα και κυρίω αν είναι λογικός μέσα σε αυτή την κρίση. Τα συζητήσαμε με τους αντιπροέδρους στην Επιτροπή των Προπολογισμών και με τον Γενικό Γραμματέα. Και θεωρώ ότι ουδέποτε δεν είχε σημειωθεί τόση ομοφωνία μεταξύ της Επιτροπής των Προπολογισμών να κάνουμε εξοικονόμηση και με την, ε, την άλλη μεριά την, ε, προτείνει ο εισηγητής Βόν και από την άλλη μεριά η διοίκηση να θέλει ε, ουσιαστικές ε, ουσιαστικές οικονομίες χωρίς να παραβλάπτει τη λειτουργία του Κοινοβουλίου. Αυτό μας το πειθούμε εδώ είναι να υπάρξει κάποιο είδου ε, νομοθεσία, νομοθεσία ε, και θα πρέπει να, η νομοθεσία αυτή να είναι ποιοτική και κυρίως να συμφωνεί ο Ευρωπαίος με αυτό. Αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε, ε, ε, λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να έχουμε αύξηση κάτω από το 2% ή τέλο πάντων άτα για το 2013. Το Προεδρείο. Έχει σαν αφετηρία την αύξηση του 3%. Και υπάρχει κάτι το οποίο μας χωρίζει ότι θέλουμε να βρούμε ένα κοινό σημείο και θα θυμάστε συνάδελφοι ότι τελικά η μέση λύση είναι καλύτερη. Και ακριβώς έτσι θα κάνουμε και θα μπορέσουμε να βρούμε την ε, εξισορρόπηση, την τέλεια των πραγμάτων. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μάνκα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο εισηγητής με μεγάλη σαφήνεια επεσήμανε τους τομεί όπου θα μπορούσε το Κοινοβούλιο να πραγματοποιήσει οικονομίες. Έδειξε ότι θα μπορούσαμε να είμαστε και αποτελεσματικότεροι στο έργο μας. Συνεργάστηκα, ε, μάλλον ε, εργάστηκα ως εισηγητής ε, για τη μελέτη του προπολογισμού του 2010 και μπορώ να πω ότι για τα θεσμικά όργανα και το Ευρωκοινοβούλιο είχαμε εντοπίσει πολλές αναποτελεσματικότητες και απώλειες πολλών χιλιάδων ευρώ ετοιμάστηκε έκθεση για το θέμα αυτό, την οποία ενέκρινε το κοινοβούλιο μας. Εκεί λέγαμε ότι χρειάζεται εσωτερικός έλεγχος. Και επίσης είχαμε συμφωνήσει να ξεκινήσει με την στήριξη της αρμόδιας γενικής διεύθυνσης ο έλεγχος αυτός. Όμως τελικά προστρέξαμε σε εξωτερικό έλεγχο και όχι σε εσωτερικό από εσωτερικό φορέα. Η αλήθεια είναι ότι αν ελέγχουμε εμεί του εαυτού μα, ποτέ δεν θα πραγματοποιήσουμε τι οικονομίε που χρειάζονται. Αυτή τη στιγμή ε, όλες οι επιχειρήσεις και οι φορείς αναζητούν ε, πόρους που μπορεί να μην είναι φανεροί. Ε, εγώ ως διαχειριστής μιας μεγάλης περιφέρειας στη χώρα μου διαπιστώνω ότι χάθηκε το 20% των εισοδημάτων μας από τις προσπάθειες εξορθολογισμού του προϋπολογισμού και νομίζω ότι εδώ έχουν γίνει πολύ καλές προτάσεις ε, στην συγκεκριμένη έκθεση. Όμως θα πρέπει να ακούσουμε και τις συμβουλές του ελεγκτικού συνεδρίου. Να δούμε πώς οι εξωτερικοί έλεγχοι θα μπορούσαν να μειώσουν και το κόστος αλλά και να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των ελέγχων μα. Ίσως αυτό να μα ε, επιτρέψει να εξοικονομήσουμε εκατομμύρια ευρώ. Ευχαριστώ για την ομιλία σα. Για 1,5 λεπτό, κύριο Χάγκλουντ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου πρώτα απ' όλα να μιλήσω με την ιδιότητά μου του συντονιστή στην ομάδα προεπολογισμών και να ευχαριστήσω το καταπληκτικό πολύ καλό εισηγητή για την πολύ καλή δουλειά του. Ε, είναι σημαντικό λοιπόν σε αυτή τη δύσκολη οικονομική περίοδο που ζούμε να υπάρχει συνένεση. Ο συνάδελφός μου κύριος Γκεμπράντη εξήγησε πολύ καλά ποια είναι η θέση της ε, ομάδας μας ε, εξετάζουμε πολύ σοβαρά όλα τα κονδύλια ε, για να μπορέσουμε να εξοικονομήσουμε κονδύλια αντί να αυξήσουμε τον προϋπολογισμό. Ε, ε, ζητήσαμε Επίσης ε, να περιστούν και δαπάνες ε, στους εξωτερικούς συνεργάτες. Αυτό το ζητάμε εδώ και πολύ καιρό. Ο κύριος Βέλε, ο Γενικός ε, Γραμματέας, έχει κάνει πολύ καλή δουλειά στο να βρίσκει εξοικονομήσεις κονδυλίων. Από τη στιγμή βέβαια που το, το ζητήσαμε. Προφανώς λοιπόν εξοικονομήσεις κονδυλίων προκύπτει μόνο εφόσον τη ζητήσει κανείς και αυτό είναι κάτι σημαντικό. Επίσης ψηφίσαμε για την ε, τροπολογία σχετικά με τη μία έδρα. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, αυτό είναι συμβολικό για κάποιους, αλλά είναι και οικονομικής φύσεως. Ε, σε δύσκολες εποχές που ζούμε, είναι σημαντικό ε, οι συνάδελφοι να τοποθετηθούν επ' αυτού του θέματος. Νομίζω ότι τα καταφέραμε αρκετά καλά και θα έχουμε πολύ καλύτερη εικόνα προς τα έξω στο μέλλον. Ευχαριστούμε τον κύριο Χάγκλουντ για ένα λεπτό. κύριος Πίτερ Βαντάλεν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε πρόεδρε, τα κράτη-μέλη ε, κάνουν ε, εξοικονόμηση κοντιλιών εδώ και χρόνια και αυτό είναι σωστό. Αλλά από ό,τι φαίνεται οι ευρωπαϊκοί θεσμοί δεν το έχουν καταλάβει αυτό. Ε, ζητούν όλο και περισσότερα χρήματα. Η έκθεση του συναντέλφου Βον επιτέλους βάζει τέλος στις σπατάλες και γι' αυτό τον συγχαίρουμε. Η έκθεση Ζητάει επίσης ε, και την ε, ανεξάρτητη εξολόγηση του προπολογισμού από εξωτερικούς ε, εμπειρογνώμονες. Εδώ δεν συμφωνώ, μάλλον από εσωτερικούς ελεγκτές. Εδώ δεν συμφωνώ, δεν μπορούμε μόνοι μας να κρίνουμε τον εαυτό μας. Πρέπει να το αναθέσουμε σε εξωτερικούς συνεργάτες. Πρόκειται για μία κοιλίδα μαύρη κοιλίδα το ότι ε, δεν ε, τεκμηριώνται οι δαπάνες ε, των ευρωβουλευτών. Τα πρέπει να τεκμηριώνται. Μετά από δική μου πρωτοβουλία το 2012 συνδέεται με κάποιες επιφυλάξεις και χαίρομαι γι' αυτό. Πρόεδρος, ο κύριος Συνάδελφοι, ε, μιλάμε εδώ για μείωση της σπατάλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο, αλλά δεν αναφέρεται αυτό που είναι η πραγματική κατασπατάληση και το γνωρίζουμε όλοι. Το να υπάρχουν δύο κοινοβουλευτικές ε, έδρες ε, κοστίζει τουλάχιστον 200 εκατομμύρια το χρόνο και σε μία θητεία ένα δις ευρώ. Νομίζω λοιπόν ότι αν το ήξεραν αυτό οι Ευρωπαίοι πολίτες θα μας έπαιρναν με τις πέτρες. Δεν μπορούμε να ζητάμε θυσίες από τους άλλους και από την άλλη εμείς να τα αυτά τα χρήματα που είναι άχρηστα είναι πεταμένα σχεδόν όλες οι πολιτικές ομάδες πρέπει να συμφωνήσουν για να δούμε κατά πόσο μπορούμε να δώσουμε μήνυμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Η ε, Προεδρία της Δανίας εκφράστηκε κατά της διπλής έδρας. Σήμερα το έκανε περίπου και ο κύριος Μόντι ε, αποφεύγοντας να απαντήσει. Δεν μπορούμε λοιπόν πλέον να αντιμετωπίζουμε αυτή την, ε, τον αναχρονιστικό εκβιασμό των Γάλλων. Ευχαριστούμε πολύ για 1,5 λεπτό. Ο κύριος Χάρτουγκ. Πρόεδρε, στις κάτω χώρες λέμε ότι δεν αρκούν τα λόγια, αλλά χρειάζονται πράξεις. Εδώ για την ώρα έχουμε ακούσει μόνο λόγια και καμία πράξη δεν έχουμε δει. Το πάγωμα των δημοσιονομικών γραμμών είναι κάτι το παράξενο, διότι τώρα έχουμε αποκτήσει περισσότερες αρμοδιότητες. Και φαίνεται ότι όλα αυτά θα κοστίσουν δισεκατομμύρια ευρώ στους πολίτες μας. Πρέπει λοιπόν να μεταρρυθμίσουμε και να αναθεωρήσουμε τον τρόπο που λειτουργούν τα θεσμικά μας όργανα. Η Επιτροπή των Περιφερειών ζητήθηκε να γνωμοδοτήσει για το θέμα αυτό, αλλά ούτε εκείνοι έκαναν κάτι τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλούνται να κάνουν και εκείνοι οικονομίες. Όμως το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν έχει αναλάβει καμία δράση, ούτε έχει κάνει καμία προσπάθεια, ε, προσπάθεια εξοικονόμησης. Υπήρξαν και άλλα στοιχεία του προπολογισμού που έχουν παγώσει στο παρελθόν, όπω τα οδημπορικά. Όμως, εδώ χρειαζόμαστε πραγματικές οικονομίες. Λόγω χάρη, το οίκο της ιστορίας κοστίζει 75 εκατομμύρια ευρώ στου πολίτε. Ποια είναι η λύση που θα εξεύρουμε. Ας δημιουργήσουμε μια ομάδα εργασίας. Ακούγεται κάπω αστείο ίσως, όμως είναι πραγματικά η κατάλληλη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση να αφήσει τα σοσιαλιστικά ιδεώδη και να σκεφτεί πραγματικά τους πολίτες. Οι πολίτες αρχίζουν να μην αντέχουν άλλο. Ευχαριστούμε. Τώρα για δύο λεπτά ο κύριος Φερνάντες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνάδελφοι, θα ήθελα σε κάθε περίπτωση να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον εισηγητή καθώς και τους κοιόδης εισηγητές για το εξαιρετικό του έργο. Νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να θυμόμαστε κάποιους αριθμούς για να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Φέτος, ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση φτάνει τα 129 εκατομμύρια ευρώ. 1% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσαμε να σημειώσουμε ότι οι προπολογισμοί και των 27 κρατών μελών είναι 44 φορέ μεγαλύτεροι από τον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωσης. Άλλο ενδιαφέρον αριθμό μεταξύ του 2000 και του 2010. Οι προπολογισμοί των κρατών αυξήθηκαν κατά 60%, ενώ ο ευρωπαϊκό προπολογισμό κατά 35%. Κατά την ίδια περίοδο, να μην ξεχνάμε ότι διαβρύθηκε κατά 12 νέα κράτη-μέλη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο προπολογισμό λοιπόν τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να γίνεται αντιληπτό ω μια μεγάλη επένδυση ε, πέραν των διοικητικών δαπανών για όλα τα θεσμικά όργανα, που καταλαμβάνουν μόνο το 6% του προπολογισμού. Οι διοικητικέ δαπάνε και οι δαπάνε λειτουργία του Ευρωκοινοβουλίου εκπροσωπούν το 1% του προπολογισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το ποσοστό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει βεβαίω να συνεχίσουμε να απαιτούμε περισσότερα και να μην εφαρμόζουμε τις αρχές οικονομίας και αυστηρότητας. Το αντίθετο. Θα πρέπει να είμαστε συνεπείς στις αρχές της εγκράτειας, της καλής διαχείρισης, της χρηστής οικονομικής διαχείρισης και στην ε, διακυβέρνησή μας και στο σχεδιασμό των προπολογισμών μας. Όπως κάναμε με το διοικητικό προπολογισμό και των άλλων θεσμικών οργάνων και του Ευρωκοινοβουλίου για τη φετινή χρονιά θα πρέπει να πετύχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή αυστηρότητα και όσο δυνατόν περισσότερε αποταμιεύσει και οικονομίε. Θα πρέπει να δαπανούμε του ελάχιστου ελάχιστους πόρου πόρους για τη λειτουργία των θεσμικών οργάνων στην περίπτωση του Κοινοβουλίου. Θα πρέπει να επιβεβαιώσουμε από την κοινοβουλευτική μα σκορπιά ότι βρισκόμαστε σε σωστή πορεία. Σα ευχαριστούμε. Για δύο λεπτά, η κυρία Γκαρτία Ζεμπάλε Ρομπέρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να αρχίσω με συγχαρητήρια προ τον κύριο Βον. Τον εισηγητή, διότι επιτέλεσε εξαιρετικό έργο, διότι εδώ μα παρουσίασε κάποιε καλύτερε γραμμέ για τον προπολισμό του Κοινοβουλίου. Και ακολουθεί τον δρόμο που χαράξαμε εδώ και κάποια χρόνια και αυτή η μέθοδο τελικά συγκεντρώνει την γενικότερη επιδοκιμασία και θα πρέπει επίση να σα πω ότι εδώ είμαστε, έχουμε ένα προπολισμό 1% μόλι πάνω από τον, τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, εάν συγκρατεί αυτός ο προπολογισμός, ε, θα, θα μπορεί να μας οδηγήσει με επιπλέον μέτρα σε συγκράτηση των εξόδων. Επίσης, μιλάμε τώρα για το τι θα κάνουμε το 2013 και ο στόχος αυτής της ε, πρώτης ψηφίσματος είναι το να έχουμε κάποιες κατευθυντήριες για τον προπολογισμό σε σχέση με το πώς θα δουλέψουμε τους αμέσως επόμενους μήνες. Και έχουμε επομένως αυτές τις προτεραιότητε για το 2013. Προτεραιότητε οι οποίε θα διακρίνονται από ευθύνη δημοσιονομική και θα μειώσουμε τα έξοδα χωρίς όμως να παραβλάψουμε το έργο ε, αυτού, αυτού του Κοινοβουλίου και έτσι θα μπορέσουμε να, να φέρουμε αυτό το πάγμα το οποίο θέλουμε στον προπολογισμό και προτείνουμε να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να μειωθούν τα έξοδα για τα ταξίδια. Και όσον αφορά τώρα τις ε, αποζημιώσεις, ε, προτείνω μέχρι το τέλος της θητείας να παγώσουν και έτσι θα πρέπει να πάμε και να κάνουμε έτσι σημαντικές οικονομίες μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επίσης. Γι' αυτό και εμείς ε, προτείνουμε ε, ε, με τρεις τρόπους να προχωρήσουμε. Πρώτα-πρώτα να έχουμε αυτή την ανεξάρτητη εκτίμηση, να συγκροτήσουμε μια ομάδα εργασίας που ασχοληθεί με αυτό εδώ στο Κοινοβούλιο, που να μελετήσει διάφορες λύσεις και τέλος ζητήθηκε από τον Γενικό Γραμματέα να κάνει μια μια τέτοια έρευνα, ούτως ώστε να μην έχουμε επικαλύψεις ενεργειών Θεωρώ επομένω ότι τα μέσα τα οποία ήδη θα ληφθούν ε, έτσι θα μας βοηθήσει να έχουμε μια καλύτερη, ε, καλύτερη διαχείριση των χρημάτων των οικονομικών μας. Ο πρόεδρος, ευχαριστώ πάρα πολύ και τώρα για 1,5 λεπτό. Η κυρία Γιάννη έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι είναι πραγματικά λυπηρό το γεγονός ε, ότι δεν μπορούμε να επιτύχουμε το αυτονόητο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δηλαδή να σταματήσει αυτό το τσίρκο των ταξιδιών ανάμεσα στις ε, έδρες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά αυτό όμως δεν μπορούμε να το αποφασίσουμε εμείς. Ε, δυστυχώς μπορούν να το αποφασίσουν μόνο οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των κρατών μελών. Και εγώ πιστεύω ότι πρέπει να καταστήσουμε πιο αποτελεσματική την εργασία μας και να προσπαθήσουμε να προβούμε σε εξοικονομήσεις κονδυλίων. Όμως αυτό όχι εις βάρος της πολυγλωσσίας. Είναι πολύ σημαντικό να βρούμε τεχνικές λύσεις οι οποίες οδηγούν στην εξοικονόμηση κονδυλίων αλλά παράλληλα και σε καλύτερη ποιότητα μετάφρασης και διερμηνίας δεν πρέπει να επιτρέψουμε την επιδίνωση των γλωσσικών υπηρεσιών. Χαίρομαι πάρα πολύ που ε, θα παγώσουν οι δαπάνες. Πρέπει όμως ε, να υπογραμμίσουμε ότι όλοι οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να επιδιώξουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Αυτό ισχύει για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, για το Συμβούλιο, για την Επιτροπή των Περιφερειών και για πολλούς άλλους. Η ε, ένταξη της ε, Κροατίας μπορεί να αποτελεί και έναυσμα για να δούμε πού μπορούμε να επιτύχουμε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Θα ήθελα το στο λόγο στον κύριο ε, Φόξ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε και θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας ε, τον κύριο Βον για τη δουλειά του. Ε, και συμφωνώ και εγώ ότι πρέπει να υπάρξει πάγωμα ε, δαπανών το 2013. Αυτή είναι η ε, πρώτη φορά που ε, δέχονται οι εργατικοί ε, και ίσως με τον τρόπο αυτό να ξεκαθαρίσουν λίγο τον κόπρο του αυγία που άφησαν φεύγοντες. Ελπίζω αυτό κύριε Βόν να το λάβουν υπόψη τους τα αφεντικά τους. Κάθε χρόνο για τα επόμενα 7 χρόνια πρέπει να υπάρξει εξοικονόμηση. Παραδείγματος χάρη ίσως οφείλουμε να καταργήσουμε την άχρηστη κοινωνική επιτροπή και την άχρηστη επιτροπή των περιφερειών. Με τον τρόπο αυτό θα εξοικονομήσουμε χρήματα των φορολογουμένων και θα περιορίσουμε την ε, γραφειοκρατία. Και να έχουμε και μία μόνα έδρα, να μην γίνεται κάθε φορά αυτό το πήγαινε έλα ανάμεσα σε Βρυξέλλες και Στρασβούργο. Κύριε Πρόεδρε, στην πατρίδα μας έχουμε λιτότητα και οι εκλογέ μας παρακολουθούν τον τρόπο που αντιδρούμε και καλό τα μέλη να στηρίξουν αυτή την έκθεση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρο η κυρία Ματέρα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, ε, βρισκόμαστε σε ένα δύσκολο οικονομικό και χρηματοπιστωτικό πλαίσιο ε, σε ολόκληρο τον κόσμο. Έχουν φανεί οι αδυναμίες πολλών κρατών μελών και πολλά εξ αυτών ζητούν από τους πολίτες τους ε, μεγάλες θυσίε για να ξεφύγουν και να ξεπεράσουν αυτή την ύφεση που δεν έχει προηγούμενο Οι γραμμές που προβλέπονται στον προϋπολογισμό καθοδηγούνται από εξοικονόμηση κονδυλίων. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι απαραίτητο να ζητήσουμε ε, περιορισμό των δαπανών, κάτι που ζήτησε ο κύριος Λεβαντόφσκι, 1,9% θα είναι η μέγιστη αύξηση των διοικητικών δαπανών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που θα πλησιάζει περίπου τον προπολογισμό τον εκτιμούμενο προπολογισμό για το 2013. Το Κοινοβούλιο οφείλει να ακολουθεί στην ίδια γραμμή όσον αφορά τις ε, δαπάνες του και για τους μισθούς ε, και για την πολιτική ακινήτων. Βεβαίως ε, να μην πέσει στον πειρασμό των λαϊκίστικων τροπολογιών. Δεν θα είναι εύκολο να απαντήσουμε σε αυτούς που έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους απέναντι στην Ευρώπη. Όμως ο προπολογισμό αυτός είναι μόνο το 2% του συνόλου των δαπανών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει λοιπόν να αποδείξουμε ότι ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε θέση να ε, συνεισφέρει ε, υπεραξία ε, και να στηρίξει επενδύσει σε εκείνε τι πολιτικέ που εντάσσονται στη συνταγή για να ξεπεράσουμε την κρίση οι απαντήσεις μας ε, πρέπει να οδεύουν προς την ανάπτυξη. Αυτός είναι ο στόχος μας και αυτό θα αποτελεί απόδειξη της αξιοπιστίας μας ε, για το 2013. Ευχαριστώ Πρόεδρε και πάλι συγχαρητήρια στον άλφο κύριο Βόν. Για τρία λεπτά ο κύριος Φέρμ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ιδιαίτερες ευχαριστίες στον κύριο Βόν, τον εισηγητή μας ο οποίος ε, έκανε μια έκθεση ιδιαίτερα σοβαρή, εξαιρετική θα έλεγα, για τον προπολογισμό του Κοινοβουλίου και των υπόλοιπων θεσμικών οργάνων. Πολύ καλά συνεργάστηκε και με τους συζητητές των υπολείπων πολιτικών ομάδων και γι' αυτό καταλήξαμε και σε συμφωνία. Αυτό αξίζει να το σημειώσει κανείς. Υπάρχει εδώ μια νέα στάση, μια νέα συμπεριφορά. Ο προπολογισμό του κοινοβουλίου, του κοινοβουλίου αυξανόταν διαρκώ χρόνο με το χρόνο. Όμω τώρα υπάρχει η γενικότερη συμφωνία ότι θα πρέπει να παγώσει ο προπολογισμό και να προβλέψουμε και την ανάγκη εξοικονομήσεων σε πολλού μεμονωμένου τομεί. Όλοι συμφωνούν ότι μπορούμε να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί στη λειτουργία μα και να δούμε και πόσο κοστίζει το λειτουργήμα των Ευρωβουλευτών. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε και τις τροπολογίες, αλλά και τι ρεκόρ εκπροσωπούν κάποιοι από τους αριθμούς. 20% ήταν ένα ποσοστό που προβλεπόταν ε, για την αύξηση των δαπανών της Επιτροπής. Τώρα έχουμε πει στο 19% 17 εκατομμύρια εξοικονόμηση δηλαδή. θα πρέπει να αναζητήσουμε την αποδοχή του κόσμου που μας παρακολουθεί, όχι μόνο επιβάλλοντας περικοπές, αλλά γεννόμενοι και πιο αποτελεσματικοί. Θα πρέπει λοιπόν οι βασικέ μα δραστηριότητε να μην χάσουν τίποτα από την ποιότητά του. Να παραμείνουμε πιστοί στο κοινοβουλευτικό μα έργο με συστηματική προσπάθεια. Με μεγάλη ικανοποίηση λοιπόν βλέπω ότι καταλήξαμε σε συμφωνία προκειμένου να δημιουργηθεί ομάδα εργασία στο Κοινοβούλιο η οποία με τη συμμετοχή εξωτερικών απειρογνωμόνων να δει που μπορούν να γίνουν οι μεγαλύτερε προσπάθειε. Τα κτίρια, την ενέργεια, την ε, συντήρηση, τα ταξιδιωτικά τους διαγωνισμούς μπορούμε πολλά εδώ να διαταχθούμε σε σχέση με το τι συμβαίνει στην υπόλοιπη, τις κρατικές δημόσιες δικήσεις. Και βεβαίως όταν σκεφτόμαστε τις υπηρεσίες διερμηνίας, μετάφρασης και ούτω καθεξής, θα πρέπει να σκεφτόμαστε πώς λειτουργούν και άλλα κοινοβούλια και άλλα κοινοβουλευτικά σώματα. Βεβαίως υπάρχει κόστος που στο κοινοβούλιο μας δεν μπορεί να συγκριθεί με τη λειτουργία άλλων κοινοβουλίων. Τα οδηπορικά, τα έξοδα διερμηνίας, Όμω θα πρέπει και η άποψη των Εθνικών Κοινοβουλίων να λαμβάνεται υπόψη. Και εδώ δεν μιλώ συντονιστή τη ομάδα μου, αλλά ω ε, Σουηδό Σοσιαλδημοκράτη. Θα πρέπει, εάν θέλουμε να γινόμαστε σεβαστοί από του συμπολίτε μα, να αξίζουμε την εμπιστοσύνη του. Να αξίζουμε την εμπιστοσύνη των φορολογουμένων. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε τα πηγενέλα μεταξύ Βρυξελών και Στρασβούργου. Απευθύνω λοιπόν έκκληση προ τι κυβερνήσει που θέλουν να σταθεροποιηθεί ο προπολογισμό Ευρωπαϊκή Ένωση να θέσουν αυτό το θέμα επιτάπητο. Εγώ σα ευχαριστώ και τώρα για δύο λεπτά ο κύριο Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρε. Χαίρομαι πάρα πολύ που σήμερα στο Στασβούργο διεξάγουμε αυτήν τη συζήτηση. Και ιδίω ε, με χαρακτήρα που συζητούμε τα σχετικά με τα κτίρια Το Στρασβούργο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι μια γέφυρα στην Ευρώπη και ακριβώς αυτό ρομαντιστεί και ο πρόεδρος Σούμανος, συνειδητής της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. Έτσι, αυτή είναι η βάση, αυτή τη διάγνωση που προς το μέλλον. Έχουμε λοιπόν ε, το κανάλι Άρτε και θα πρέπει να είμαστε υπερήφανοι για αυτό το πολιτιστικό κανάλι. Ε, θα πρέπει ε, να φτιάξουμε και ένα στούντιο εδώ στο Κοινοβούλιο γιατί εκεί μπορεί να συναντιέται η Ευρώπη και να βάζει τα θεμέλια σε σημαντικά θέματα. Στην τροπολογία 2 γίνεται λόγος για μία και μόνο έδρα. Μα κυρίε και κύριοι έχουμε μία και μόνο έδρα. Αυτή η μία έδρα είναι το Στρασβούργο και νομίζω ότι πρέπει να παραμείνουμε Μένουμε πιστοί στις ε, συμφωνίες που έχουμε συνάψει. Αυτό είναι αυτονόητο. Τροπολογία υπαρτιμών 4. Συζητάμε για τον οίκο της ε, ευρωπαϊκής ιστορίας. Νομίζω ότι είναι καθήκον μας να δείξουμε στους ε, νέους μας πόσο σημαντικό είναι να διεκδικούμε κάθε ημέρα την ειρήνη. Και αυτό πρέπει να το τεκμηριώνουμε. Έχουμε κέντρο επισκεπτών ε, που, ε, το οποίο επισκέπτονται πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι το χρόνο. Οι άνθρωποι επιθυμούν να γνωρίζουν ε, ποια ήταν ακριβώς η ιστορία της Ευρώπης και για να το πετύχουμε αυτό χρειαζόμαστε και ισχυρά πολιτικά κόμματα. οφείλουμε να έχουμε ένα μέτωπο απέναντι στους εθνικισμούς. Χρειαζόμαστε μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση, ισχυρά κόμματα και αυτά βεβαίως πρέπει κάπως να χρηματοδοτούνται. Εφόσον ε, λοιπόν στην τροπολογία υπαριθμών 6 μιλάμε για την εκπροσώπηση, ναι και οι επισκέπτες ε, έχουν ε, δικαίωμα συνοδείας να τους συμπεριφερόμαστε σωστά. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι αυτή η τροπολογία είναι πολύ σημαντική για αύριο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε λέει ο Πρόεδρος και θα ήθελα τώρα να δώσω δύο λεπτά στον κύριο Σταυρακάκη παρακαλώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον εισηγητή μα για την έκθεσή του και την εξαιρετική δουλειά του. Για ακόμα μια χρονιά η συζήτηση για την κατάρτιση των κατευθυντήριων γραμμών για το διοικητικό προπολογισμό των θεσμικών οργάνων τη Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνει η χώρα με την οικονομική και κοινωνική κρίση να βάζει σε σκληρή δοκιμασία του προπολογισμού όλων των χωρών παντού στην ευρωπαϊκή ένωση οι προπολογισμοί καταρτίζονται στη βάση εξορθολογισμού των δημοσιονομικών δαπανών και σκληρών οικονομικών μέτρων σε πολλού τομεί τη οικονομία. σε αυτή την κατεύθυνση υποστηρίζω τη θέση του εισηγητή για την ανάγκη αποφυγή περιττών και μη άμεσα αναγκαίων εξόδων με σαφή καθορισμό των προτεραιοτήτων και όπου είναι δυνατό και χρήσιμο με ανακατανομέ δαπανών έτσι ώστε να επιτευχθεί ο εξορθολογισμό του διοικητικού προπολογισμού των θεσμικών αυτών οργάνων ωστόσο όπω και ο συγητή, έτσι και εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι ο εξορθολογισμό των διοικητικών δαπανών πρέπει να λάβει υπόψη του την ανάγκη να τηρηθούν οι νομικέ δεσμεύσει τη ευρωπαϊκή ένωση όπω η προσχώρηση τη κροατία καθώ και η ανάγκη διατήρηση μια αποτελεσματική διοίκηση που θα μπορεί να ανταπεξέλθεται στι αυξημένε αρμοδιότητε του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου όπω απορρέουν από τη συνθήκη τη λισαβόνα. Λοιπόν, για ένα μισή λεπτό ο κύριος Σον ε, Καλή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Βον για την πάρα πολύ καλή δουλειά που έκανε σε αυτό το τόσο ε, σημαντικό θέμα. Κυρίως ε, τα μέσα ενημέρωσης ε, ε, στρέφουν το βλέμμα στους πολιτικούς και στις δαπάνες. Αυτό δεν είναι από μόνο του κακό. Είναι μια ευκαιρία και μόνοι μας να εξετάζουμε τα του οίκου μας. Και γι' αυτό δεν έχω καμία αντίρρηση απέναντι στην πρόταση ότι θα πρέπει εξωτερική εμπειρογνώμονες να ελέγξουν τις ε, δραστηριότητές μας. Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε και να υπεραμεινθούμε των ε, δαπανών μας ε, και επίσης θα μπορούμε ίσως να εξετάσουμε και το μίσο που θα μπορούσαμε να κάνουμε εξοικονόμηση κονδυλίων. Μέχρι τώρα πολλοί μίλησαν για την μία και μόνο έδρα του Κοινοβουλίου. το να συζητάζουμε, συνεδριάζουμε μία φορά το μήνα εδώ στο Στρασβούργο, πολλοί πολίτες δεν το κατανοούν αυτό. Είναι λοιπόν απαραίτητο να συζητηθεί το θέμα και ίσως να καταλήξουμε σε μία συμφωνία με τους Γάλλους για το Στρασβούργο. Ε, ίσως μπορούμε να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα. Και οι άλλες επιτροπές, η Επιτροπή των Περιφερειών πρέπει να την εξετάσουμε. Ε, ένας εξωτερικός έλεγχος, κατά την άποψή μου, είναι ευπρόσδεκτος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Μετεκάλη, δέχεστε ε, μπλε κάρτα από τον κύριο Ρούμπιχ. Κύριε Ρούμπιχ, έχετε το λόγο. Σύνολο Κέλλη, σας ευχαριστώ διότι θίξατε τις δαπάνες των Ευρωβουλευτών. Πιστεύετε ότι οι βουλευτές που συζητάνε εδώ για την μείωση των ε, φάπαξ ε, ποσών. Ε, πιστεύετε ότι κάθε βουλευτής είναι μόνος του υπεύθυνο για το πόσα χρήματα θα δαπανά. Δεν χρειάζεται να υπάρχει ανωτατόριο. Μόνος του μπορεί να ρυθμίζει τις δαπάνες του και στις, στους μισθούς του. Αν θεωρεί ότι παίρνει πάρα πολλά χρήματα, να δίνει δωρεές σε ανέργους, ανθρώπους που έχουν ανάγκη και αυτά να τα ε, πούμε προς την ε, κοινή γνώμη. Πιστεύετε ότι αυτός είναι ένας ε, σωστός δρόμος, δηλαδή κάθε ευρωβουλευτή να αναλαμβάνει μόνος την πρωτοβουλία. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ρουμπίκ. Βεβαίω εναπόκειται στα κράτη-μέλη να αποφασίσουν τι θα κάνουν. Αλλά κοιτάξτε, το, να αποφασίσουμε για τον εξωτερικό έλεγχο, αυτό είναι ο πλέον αντικειμενικό τρόπο. Ο Σέξπιρ είπε ότι δεν βλέπουμε τα πράγματα με αντικειμενικά μάτια. Και ίσως ε, θα μπορούσαμε λοιπόν να λάβουμε κάποια μέτρα αν αυτό κριθεί απαραίτητο. Για δύο λεπτά ο κύριος Ολένιτσακ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την ε, πολύ πλήρη και ευφυή έκθεση που μα υπέβαλε μετά την θέση σε ισχύ τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε νέε προκλήσει. Η ποιότητα τη δουλειά μα, το μέλλον θα καθορίσει το μέλλον τη ε, Ευρώπη των Ευρωπαίων πολιτών. Υπάρχουν μεταρρυθμίσεις στην κοινή αγροτική πολιτική και την πολιτική συνοχή που θα είναι καθοριστική σημασία, αλλά και σε άλλους τομεί όπου να είμαστε αποτελεσματικοί. Πρέπει να είμαστε να έχουμε συνείδηση της επαγγελματικής μας υποχρέωσης, της επαγγελματισμού μας και να είμαστε υπεύθυνοι για χρηστή διαχείριση των πόρων και για το προσωπικό ε, την ε, πολιτική προσωπικού. Υπάρχει κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γι' αυτό πρέπει να επιδείξουμε εδώ και αλληλεγγύη, διάθεση αλληλεγγύης, γιατί υπάρχουν πολίτες που πρέπει να κάνουν οικονομίες ε, καθημερινά, όχι μόνο οι Έλληνες, αλλά και οι Πολωνοί και οι πολίτες άλλων χωρών. Θα ήμουν λοιπόν υπέρ του παγώματος του προπολογισμού του Ευρωκοινοβουλίου. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να αναζητήσουμε εύστοχε λύσει, ακόμη αποτελεσματικότερε. Σήμερα ακούσαμε να αναφέρεται το θέμα τη έδρα του Ευρωκοινοβουλίου, τη έδρα του Στρασβούργου. Αυτό είναι κάτι που εμεί το θεωρούμε ακατανόητο. Ακατανόητο για εκατομμύρια Ευρωπαίου. Ευρωπαίου που δεν καταλαβαίνουν γιατί το Ευρωκοινοβούλιο έχει δύο έδρε. Θα πρέπει να μπει κάποια τάξη στο ζήτημα αυτό. Θα πρέπει να πάυσει αυτή η γελία κατάσταση. Εγώ είμαι υπέρ τη μία και μόνη έδρα του Ευρωκοινοβουλίου. Μία έδρα και μάλιστα στι Βρυξέλλε. Ξέρετε πόσα εκατομμύρια ευρώ εξοικονόμηση θα σήμαινε κάτι τέτοιο. Για ένα λεπτό, ο κύριος Κοάλ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή για την έκθεση τελική ανάλυση όμως ε, δεν βοηθάει σε τίποτα γιατί όλα αυτά συρρυκνώνονται σε τρεις λέξεις. Οικονομία, οικονομία, οικονομία. Αν θέλουμε να ε, δώσουμε το καλό παράδειγμα στους Ευρωπαίους μόνοι μας ε, πρέπει να κάνουμε οικονομία, να δώσουμε όπως είπα το καλό παράδειγμα. Εσείς θα εμπιστεύαστε κάποιον που δεν ρυθμίζει του οίκου τους εδώ πρέπει να ξεκινήσουμε. Δαπανάμε πάρα πολλά χρήματα για προπαγάνδα, για ε, δραστηριότητε και συμφωνώ με τον κύριο Ρούμπιχ ότι πρέπει πράγματι ε, να χρηματοδοτήσουμε τον οίκο της Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Αλλά καλύτερη διαφήμιση για μας είναι αν περιορίσουμε τις ε, δαπάνες μας. Έτσι θα δίναμε και το καλό παράδειγμα. Πρόεδρος, Φτάνουμε τώρα στη διαδικασία του Catch the Eye και πρώτη θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Μπασέσκου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρόεδρε, αυτή τη στιγμή τα κράτη-μέλη είναι πάρα πολύ σημαντικέ δημιουργικέ δυσκολίε, οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να κυριαρχήσει η, η μεσομική Θα πρέπει ε, τα θεσμικά όργανα να είναι υπεύθυνα και να έχουν πολιτική λιτότητα. Σε αυτή τη στιγμή οι διοικητικέ δαπάνε είναι περί τα 5,8% του συνολικού προπολογισμού της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να κάνουμε περαιτέρω περικοπές και εξοικονομήσεις και θα πρέπει να δούμε πού ε, δεν έχουμε αποτελεσματικότητα στα κονδύλια, πού έχουμε επικαλύψεις. Επίσης θα πρέπει να αναλύσουμε με τι δυνατότητες έχουμε, τι, έχουμε για τις εξοικονομήσεις και έτσι να έχουμε ένα σύστημα management το οποίο βασίζεται στη γνώση. Θα πρέπει να ακολουθήσουμε όλε τι βασικέ αρχέ του άρθρου 27 για την χρηστή διαχείριση όσον αφορά τον δημιουργικό κανονισμό και οπότε στα πλαίσια αυτά θεωρώ ότι θα πρέπει οι προπολογισμοί των θεσμικών οργάνων να είναι αποτελεσματικοί και λογικοί. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρο. Ο επόμενο ομιλητή τώρα είναι ο κύριο Κοσλόφσκι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρε. Νομίζω ότι στα, στη συγκυρία αυτή που έχουμε την οικονομική κρίση και το, το, το πόσο α, βαραίνει το κρατικό χρέος θα πρέπει τα κρατημέλη να επιδείξουν ε, υπευθυνότητα αλλά και δημοσιονομική πειθαρχία. Συμφωνώ με τον εισηγητή ότι στο άμεσο μέλλον θα πρέπει να έχουμε ρεαλιστικό προϋπολογισμό. Θα πρέπει να κάνουμε εξοικονόμηση δαπανών. Θα πρέπει να παγώσουμε κάποιες δαπάνες όπως τα των ταξιτίων. Το 2013 επίσης ε, θα είναι δύσκολη χρονιά δεδομένης καταστάσεως φέτος. Οπότε θα πρέπει κατά αυτή την ε, ε, θητεία να περιοριστούμε και όσον αφορά την πολιτική των κτηρίων. Νομίζω ότι και το Προεδρείο θα πρέπει να συνεχιστεί με την ε, πλευρά των Προπορισμών, τόσο ώστε να προχωρήσουμε σε κάποιε προτάσει ουσιαστικέ. Κύριο Φερέτρο, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα πρέπει εδώ να προσπαθήσουμε να κάνουμε οικονομίε στο επίπεδο όλων των θεσμικών οργάνων τη Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωκοινοβουλίου. Να μην ξεχνάμε εδώ τι μέρημνε που έχουμε σε σχέση με την αρχή τη πολυγλωσία Υπάρχουν ανεπάρκειες στις υπηρεσίες διερμηνείας και μετάφρασης, οι οποίες θέτουν εν αμφιβόλο και απειλούν την αποτελεσματική μας εργασία σε πολλές περιπτώσεις. Οι τροπολογίες αυτής της έκθεσης λόγου χάρη, όπως την Επιτροπή Προπολογισμών, θα μπορούσαν να γίνουν αποδεκτές μόνο στα αγγλικά. Αυτό σημαίνει διακριτική μεταχείριση των βουλευτών άσχετα με την εθνική τους καταγωγή. Πρέπει λοιπόν οι περικοπέ τη υπηρεσία διερμηνία ε, μπορεί να επηρεάσουν οι περικοπέ αυτέ την αποτελεσματική μα λειτουργία. Και απειλούνται και εργαζόμενοι απαραίτητοι για την ε, αποτελεσματική ε, και την ποιοτική εργασία του σώματο αυτού. Για του εργαζόμενου λοιπόν στι υπηρεσίε τη διερμηνία και τη μετάφραση δεν θέλουμε καθόλου να απειλούνται τα δικαιώματα και η εργασία του. Ο κύριο Σιλβέστρη η λιτότητα για τις διοικητικές δαπάνες και τις επενδύσεις για να ε, ευνοηθεί η ανάπτυξη αυτές είναι οι λέξεις κλειδιά της κατευθυντηρίων γραμμών ε, για τον προπολογισμό του 2013. Εδώ λοιπόν θέλω να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Βόν για το έργο του διότι έδειξε για μεγάλη προθυμία και μεγάλη ελαστικότητα και διαλλακτικότητα για να συνεννοηθούμε. Στου καιρού αυτού τη οικονομική κρίση θα πρέπει να υψώσει τη φωνή τη η Ευρώπη. Χρειάζεται περισσότερη Ευρώπη, χρειάζεται οικονομική διακυβέρνηση τη Ευρώπη ισχυρή και θα πρέπει η Ευρώπη να αναλάβει το ρόλο τη δίπλα στα κράτη-μέλη. Όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτε σε όλα τα κράτη-μέλη να καταλάβουν ποια είναι η παρουσία τη Ευρώπη, πώ μπορεί να στηρίξει την ανάπτυξη. Πρέπει να γίνουν επιλογέ για τον προπολογισμό και θα πρέπει να έχουμε μια συγκεκριμένη στρατηγική για την ανάπτυξη ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για τα μεμονωμένα κάτι μέλη. Οι περικοπέ όμω, αργά ή γρήγορα, θα πρέπει να μα απασχολήσει ποια θα είναι η δαπάνη των δαπανών. Ποιε είναι αυτέ που περισσότερο αναμένουν οι πολίτε. Ποιοι είναι αυτοί που θα, ε, ποιες είναι οι δαπάνες που θα επιτρέψουν στους πολίτες να έχουν περισσότερη ε, εμπιστοσύνη στους Ευρωπαίους πολίτες. Δεν μπορούν οι πολίτες να καταλάβουν ακόμα γιατί έχουμε δύο έδρες. Ευχαριστούμε κυρία Σινκλέρ. Σας ευχαριστώ και συγχαρητήρια στον κύριο Βόν για την έκθεση και επίσης τον Επενό που θέλει να γίνει ο Κινκένι του 21ου αιώνα. Ο πρωτοπόρος δηλαδή. Δεν ήθελα να είναι πρωτοπόρος, αλλά τη συγκράτηση των εξόδων. Θέλουμε εξυγίανση των ημισονομικών. Όμως δεν το θέλει αυτό στην πραγματικότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλει περικοπές. Θέλει ουσιαστικά με την άτα να αυξήσει τα έξοδα. Θα έπρεπε να γίνουν περικοπές, να εξοικονομήσουμε δηλαδή τα χρήματα των φορολογουμένων μέσω των ανεξαρτήτων εμπειρογνώμων. Έχετε τόσα 4-5 καταστάρια μέσα σε αποζημίωση στους βουλευτές και είναι αυτοί οι βουλευτές οι οποίοι την Παρασκευή υπογράφουν ότι βρίσκονται εδώ, ενώ δεν, εδώ δεν κάνουμε τίποτα την Παρασκευή. Αυτό είναι κλοπή. Πρέπει να σταματήσει. Το ίδιο ισχύει και για τα έξοδα των γραφείων. 50% περικοπή, όχι πέρα 90%. Να γίνει έλεγχος από ανεξάρτητου ελεγκτές. Όλο αυτό είναι διασπάθηση τερατώδης των χρημάτων φορολογουμένων. Ευχαριστώ ο τελευταίος ομιλητής ο κύριος Ρούμπιχ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, σε αυτή τη συζήτηση, από αυτή τη συζήτηση προέκυψε ότι οι πολίτες έχουν δικαίωμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μαθαίνουν περισσότερα το τι ακριβώς κάνουμε εδώ, το τι μπορούν να τους προσφέρουν οι θεσμοί. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ ε, λέω ότι πρέπει να ενισχύσουμε την εικόνα μας προς τα έξω. Αυτό είναι σημαντικό για την κοινή γνώμη και όλα αυτά βέβαια πρέπει να λέγονται σε όλε τι γλώσσε. Γι' αυτό είναι και τόσο σημαντική η διερμηνή μα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το μόνο κοινοβούλιο του κόσμου ε, το οποίο έχει τη δυνατότητα να συνεννοείται με πολλέ γλώσσε. Και κατόπιν τούτου στον προπολογισμό είναι καθοριστική σημασία τα πολιτικά κόμματα και οι ευρωβουλευτέ να δραστηριοποιηθούν ακόμα περισσότερο για να εξηγήσουν την δουλειά της Ευρώπης για την ειρήνη. Να δείξουν επίσης ότι εργάζονται αποτελεσματικά, ότι δεν είναι όλοι οι ευρωβουλευτές οι ίδιοι και αυτό νομίζω φάνηκε από τη σημερινή συζήτηση. Uh, it's a blue card. Μπλε κάρτα, διαδικαστικό παρακαλώ. Πρόεδρε, στην προηγούμενη συζήτηση για τα δικαιώματα μου είχατε δώσει χρόνο και είχα και μπλε κάρτα, όμω εσεί μου λέτε να μην χρησιμοποιήσω για δεύτερη φορά την μπλε κάρτα. Αλλά και για το ΚΑΤΣΔΙ μου έδωσε ο μιλητή την άδεια να μιλήσω και στο ΕΛΚ επίση. Είχαμε επίση διάφορου οι οποίοι πήραν για δεύτερη φορά. Θα πρέπει εδώ να έχουμε ισότητα στη συζήτηση. Και αφού θέλουμε να δώσουμε το πράγμα στον εξωκόσμο, πρώτα-πρώτα την έχουμε την ισότητα στα του οίκου μα κυρία Σινκλέρ. Ε, Θα ήθελα να σας πω ότι όλοι είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν την άποψή τους και εσείς την είχατε αυτή την ευκαιρία και δεν νομίζω ότι παραβιάσαμε το καταστατικό. Και τώρα ε, το λόγο έχει ο κύριος Βον. Κύριε Βον, έχετε το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τους σκιώδη ηγητές και όλους τους συναδέλφους που μίλησαν σήμερα το απόγευμα. Από ό,τι φαίνεται υπάρχει ευρεία συνένεση στο ότι πράγματι ε, πρέπει να κάνουμε οικονομίε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να έχουμε περιορισμένο ε, προπολογισμό. Και είμαι σίγουρο ότι ο Γενικός Γραμματέας παρακολουθεί τη συζήτηση από το εσωτερικό δίκτυο. Ε, Εξοικονομίες βέβαια πρέπει να ε, διευκρινιστούν. Σήμερα είδαμε ότι υπάρχει διάσταση απόψεων για την μία και μόνο έδρα, ε, για το κόστος μετάφρασης, για τον οίκο της ιστορίας. Αυτές είναι διαφορετικές απόψεις ανάμεσα στους συναδέλφους. Όπως επίσης διάσταση απόψεων και για το ρόλο της ομάδας εργασίας ε, που σας πρότεινα. Πρέπει λοιπόν να είμαστε όσο πιο ευέλικτοι γίνεται. Σε επίπεδο ομάδας εργασίας θα εξετάσουμε τις λεπτομέρειες και θα τις επιλύσουμε. Στόχος είναι να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στις απόψεις όλων των συναντέλφων. Και σε τελική ανάλυση στόχος είναι να έχουμε ένα όσο πιο περιορισμένο προϋπολογισμό γίνεται, παράλληλα όμως να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστούμε κύριε Βόν. Έκλεισε η συζήτηση και η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο στις 12. Χαίρετε. Τι θέλετε εσείς, διαδικαστικό? εκτός μικροφώνου. Λυπάμαι πάρα πολύ. Ο μιλητής ε, μιλάει εκτός μικροφώνου. Κοιτάξτε, διαδικαστικό. Μιλάμε σε ένα κενό. Δεν έχουμε εδώ παρόντα ούτε το Γενικό Γραμματέα, ούτε τους αρμόδιους αντιπρόεδρους του Κοινοβουλίου αρμόδιους για τον προπολογισμό. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας στις επόμενες συζητήσεις που θα λάβουν χώρα, να είναι παρόντες εδώ και οι τρεις που προανέφερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συμφωνώ απόλυτα επ' αυτού μαζί σας όταν πράγματι συζητάμε τόσο σημαντικά θέματα όπως είναι ο προϋπολογισμός, ε, αυτοί που είναι αρμόδιοι, τόντι, θα πρέπει να είναι παρόντες. Ε, συμφωνώ απόλυτα με τα σχόλιά σας και θα το δείξω θέμα στην συνεδρία του Προεδρείου. Καλό σας βράδυ. Uh, denní 9 Η συνεδρίαση λήγει ως αύριο, μάλλον ως το βράδυ στις 9.